Good afternoon, ladies. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, παρακαλώ. Και καταρχήν ε, ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη ή με το υπάρχουν σχόλια. Όχι από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστώ. Άρα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις ε, της Προέδρου δεν υπάρχουν, για σήμερα τουλάχιστον. Ίσως αργότερα προκύψουν. Περάμε στο τρίτο σημείο της ημερήσης διάταξης, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων για τις εδαφικές τυπολογίες. Μαζί με τους ε, ε, αρμόδιους για τη διαμόρφωση πολιτικής, η Eurostat έχει ξεκινήσει μελέτες προκειμένου να ε, δημοσιεύει στα, στατιστικές με βάση τις ε, δαφικές τυπολογίες όπως θέματα ε, αστικών αγροτικών περιοχών παράκτων και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμής ο κανονισμός ΝΑΤΣ δεν κάλυπτε αυτές τις περιφερειακές τυπολογίες, τις εδαφικές τυπολογίες. Και αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι τεχνικής φύσης και στόχο έχει να αναγνωρίσει νομικά τις ε, τυπολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται. Ζητήσαμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει τους τα βασικά στοιχεία της πρότασής της ε, και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια εισαγωγή που θα μας κάνει ο αρμόδιος εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν θα έχουμε συζήτηση με τους και και την εισηγήτρια που είναι υποφαινόμενη. Ξεκινάμε λοιπόν με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Νούλε. Ή μήπως υπάρχουν αλλαγές εσείς είστε. Ναι. Δεν λέγομαι όμως Νούλε, αλλά Γκούντε Σέφερ. Είμαι αρμόδιος θυματάρχης για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας να παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή για να γίνει διεξοδική συζήτηση προκειμένου να γίνει αποδεκτή η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ και πολλά χρόνια, για να σας εξηγήσω το ιστορικό υπόβαθρο, ασχολούμαστε με τα θέματα της τυπολογίας, γιατί όπως θα φαντάζεστε δεν είναι εύκολο να, να λαμβάνουμε υπόψη τις ε, επιμέρους περιοχές για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά και για θέματα πολιτικής μιλούμε για πολλά είδη περιφερειών και περιοχών. Ε, αστικές, αγροτικές, παράκτιες, θαλάσσιες και ούτω καθεξής. Και για στατιστικούς λόγους χρειαζόμαστε κάποιες τυπολογίες ε, για να κάνουμε στις στατιστικές μας διαφοροποίηση μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών στις πόλεις για παράδειγμα ή στις αστικές περιφέρειες και μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών. Χρησιμοποιούμε εδώ και καιρό αυτές τις τυπολογίες και τις έχουμε ε, εμπεδώσει, εδραιώσει και ενοποιήσει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα στην πράξη χρησιμοποιούνται από πολλές ε, γενικές διευθύνσεις πολιτικής, αλλά και γενικώ αυτές οι τυπολογίες. Και όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, ουσιαστικά θα προσθεθούν στον κανονισμό ΝΑΤΣ Τη κοινή ονοματολογία εδαφικών στατιστικών ομάδων, που είναι ένα ευρεωμένο σύστημα που εξυπηρετεί όχι μόνο στατιστικούς σκοπούς αλλά και πολιτικούς. Και χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των περιφερειών και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυπολογίες που τώρα προσπαθούμε να ενοποιήσουμε είναι αυτές που χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια ολόκληρα σε πολλούς κλάδους και για πολλούς σκοπούς. Έχουμε περιοριστεί σε, μερικούς, σε μερικές τέτοιες τυπολογίες προς το παρόν, αλλά θα εξετάσουμε και άλλες στο μέλλον. Ίσως χρειαστούν κάποιες τροπολογίες στη συνέχεια, αλλά προσπαθούμε πρώτα να αποκομίσουμε κάποια εμπειρία από τη χρήση των ε, φυσταμένων τυπολογιών και έχουμε επαφή με εμπειρογνώμονε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη ώστε να δράσουμε περαιτέρω και να ενοποιήσουμε τέτοιου είδους ε, τυπολογίε που χρησιμοποιούμε εδαφικές. Και επίσης πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση τέτοιων τυπολογιών και θα συμβάλλει στην ε, αποσαφήνιση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των ε, ευρωπαϊκών περιοχών και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση, ε, στη χάραξη ε, και εφαρμογή πραγματικά αποτελεσματικών πολιτικών στις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τώρα. Θέλει το λόγο ο κύριος Μίλλερ, η Νούλεν. Εγώ νομίζω ότι οι πιο βασικές πτυχές της πρότασης ε, δεν διαφοροποιούνται πολύ από αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε και τώρα, απλά έχουμε ομαδοποιημένα πλέον στοιχεία ανάλογα με τις αστικές περιοχές, ε, τις αγροτικές περιοχές. Ε, θέλουμε την εναρμονισμένη εφαρμογή αυτών των τυπολογιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γενικέ διευθύνσει όλες για το ίδιο πράγμα και να μα κατανοούν και τα κράτη-μέλη. ...όσα χρησιμοποιεί παρόμοια τυπολογία με αυτούς επίσης συνομιλούμε συνεχώς και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έχουμε επίσης ένα project για έναν εναρμονισμένο ορισμό των πόλεων. Και αυτό πρέπει να το λέω υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την απόφαση των συντονιστών να ακολουθηθεί η επιστευμένη διαδικασία για το θέμα αυτό. Εξού είμαι εγώ η συγγήτρια και θα ήθελα να πω δύο, λόγια για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η πρόταση έχει ως στόχο να οριστούν σαφέστερα ορισμένες γεωγραφικές ε, μονάδες για στατιστικούς σκοπούς. Οι ορισμοί αυτοί ανεπτύχθησαν σε συνεργασία με τον ΩΣΑ και έτσι έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πιο διεθνές πλαίσιο. Υπάρχουν επίσης ε, κάποιες ονοματολογίες σε επίπεδο πόλεων, δηλαδή ε, λειτουργική μετροπολιτική περιοχή, πόλη και ευρύτερη αστική περιοχή. Έχουμε κάποια project συλλογή στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα διευκολυνθούν από αυτή την νέα ε, ονοματολογία. Υπάρχουν ειδικέ προσπάθειες ιδιαίτερε προσπάθειε για την πρόθεση του αστικού θεματολογίου. Έξω και είναι πολύ σημαντικό η στατιστική βάση να υπάρχει ώστε να καλύπτονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τις πόλεις και την αστική διάσταση και την ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση θα επιτρέψει την ομαδοποίηση των δεδομένων βάσει των τυπολογιών, παράδειγμα ΑΕΠ στις ε, περιοχές υπαίθρου και στις αστικές περιοχές. Θα μπορούσε να γίνει σύγκριση. Η, απασχόληση, η, η αστικοποίηση, ο βαθμός αστικοποίησης. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για τις αστικές περιοχές και για την Ήπεθρο. Επίσης θέλουμε να έχουμε βασικούς ορισμούς και στατιστικά κριτήρια για τις διάφορες εδαφικές μονάδες και τυπολογίες ώστε να εφαρμόζονται ομοιόμορφα και εναρμονισμένα. Να χρησιμοποιούνται δε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Και η πρόταση επίση περιλαμβάνει διατάξει. που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Κομισιόν να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξης δυνάμει του άρθρου 290 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιημένο κανονισμό θα επιτρέψει τη θα δώσει τη δυνατότητα με αυτή την εναρμονισμένη ονοματολογία να γίνονται συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να στοχεύσει καλύτερα τις πολιτικές της. Η πρόταση περιλαμβάνει κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για ορισμένες από τις συγκεκριμένες πολιτικές ε, που μας ενδιαφέρουν στην δική μας Επιτροπή, ιδίως ό,τι αφορά τις αστικές περιοχές και περιφέρειες, την Ήπεθρο, αλλά και τις διαφορές μεταξύ τους. Στηρίζω προσωπικά ως εισηγήτρια λοιπόν την πρόταση και νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την επιλογή σαν διαδικασία μετά τις εξηγήσεις που ακούσαμε. Ε, υπάρχουν σχόλια από τους ε, σκιώδεις ενδεχομένως ή από άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κυρία Μάλετιτς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλει το λόγο ή δεν το θέλετε. Α, δεν το θέλετε. Η κυρία Καλ δεν είναι εδώ, Μαρζέ δεν είναι εδώ, Ροπέ δεν είναι εδώ. Ουδής παρόν. Άρα δεν υπάρχουν ερωτήσει. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Ή μήπω υπάρχουν ερωτήσει. Δεν υπάρχουν ερωτήσει. Ευχαριστώ και τους δύο κυρίους και μπορούμε να συνεχίσουμε με βάση αυτή τη διαδικασία που έχει επιλεγεί. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησιά διάταξη, που είναι η παρουσίαση του εγγράφου εργασία των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την προστέμενη αξία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Ουσιαστικά εννοούμε προϋποθέσεις ε, με στόχο το πλαίσιο πολιτικής στα κράτη-μέλη και στο θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο να προωθήσει πιο αποτελεσματικές αποδοτικές δημόσιες δαπάνες. Οι περισσότερες εκ των πατέρων ε, έχουν εκπληρωθεί από την έναρξη της ε, παρούσας περίοδου προγραμματισμού και υπάρχουν και σχέδια δράση ώστε να έχουμε ε, καλύψει και τις υπόλοιπες. Υποτίθεται ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει στα τέλη του 2016, παραμένουν όμως κάποιες εκ των προτέρων αρεσιμότητες που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Θα δώσω ως ήθιστε το λόγο καταρχά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει την αρχική παρουσίαση. 15 λεπτά το πολύ παρακαλώ και εν συνεχεία τα μέλη της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής Υποθέσεων θα πάρουν το λόγο για τις ερωτήσεις τους. Ο κύριος Γκραντ, εξ Κομισιόν, για να μας πει τα περί των προτέρων ερησιμοτήτων σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, η οποία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να, της ε, δώσει, να σας δώσει ε, μία έποψη γενική, σύντομη, των εκ των προτήτων ερασιμοτήτων, ε, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το εργαστήριο που έλαβε χώρα σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο τον μήνα Νοέμβριο. Επομένως δεν έχω πολλά πολλά να σας μάθω σχετικά με το θέμα θέμα αυτό. Θα μιλήσω ε, για τα ε, κύρια ε, ωφέλη τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, τα μαθήματα, τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει και αυτά θα τα περιγράψω εν συντομία, τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία έχουμε αποκομίσει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, να πω τα εξής αυτό το έγγραφο εργασίας βασίζεται στην εμπειρία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα ε, και στις επαφές ε, με τις ε, διαχειριστικές αρχές. Όπως είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία των εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων έχουν ήδη καλυφθεί. Έχουμε ε, λοιπόν, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στην εργασία μας με τις διαχειριστικές αρχές ότι τα πράγματα πάνε καλά. Επίσης, στη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού έχουμε ξεκινήσει μία μελέτη σχετικά με την υλοποίηση των ερεσιμοτήτων που καλύπτουν όλες αυτές τις ειδικέ διατάξεις. Όπως γνωρίζετε, κυρία Πρόεδρε, ε, οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ε, αποτελούν ε, ένα σημαντικό στοιχείο μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Ο στόχος βεβαίως είναι να υλοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν 40 εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και 36 γενικά και 36 οι οποίες αναφέρονται στην πολιτική συνοχή. Δεν θα αναφερθώ βεβαίως ε, αναλυτικά σε όλες. Ε, περίπου 75% ε, έχουν ήδη καλυφθεί και περίπου 100 προγράμματα δράσης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πρώτο προγραμματισμό έχουν ολοκληρωθεί κατά 86% όσον αφορά τις εκ των ερεσιμότητες. Βεβαίως ε, τα πράγματα δεν είναι ε, ε, τελικά ακόμα και τελειωτικά, αλλά μέχρι τον Αύγουστο του 2017 έχουν την δυνατότητα τα κράτη-μέρη να ολοκληρώσουν τα στοιχεία τους όσον αφορά τις, όσον αφορά τις προϋποθέσεις. Ιούνιο του 2017 για τα προγράμματα και Αύγουστο του 2017 όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Ε, ε, ε, βεβαίως αν μέχρι το τέλος αυτών των ημερομηνιών δεν έχουν καλυφθεί ή εκ των προτέρων θα ληφθούν μέτρα. Έχουμε όσον αφορά τα είδη των οφειλημάτων έχουμε πέντε διαφορετικούς τύπους. Το πρώτο αφορά τη γενική βελτίωση του περιβάλλοντος επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο αφορά την υποστήριξη διαφορετικών διαρθρωτικών αλλαγών και την υλοποίηση των ειδικών ε, ε, συστάσεων ε, αναχώρα. Έχουμε επίσης την βοήθεια όσον αφορά την μεταβίβαση του κεκτημένου, όσον αφορά την χρήση των ταμείων συνοχής και τέλος όσον αφορά την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και του συντονισμού. Αυτά ήθελα να πω ε, ε, πριν προχωρήσω ε, στην περαιτέρω ανάλυση. Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια συμπεράσματα της ανάλυσης όσον αφορά την πλήρωση και την κάλυψη των εκτοπροτέρων ερεσιμοτήτων είναι η εξή. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εκτοπροτέρων ερεσιμότητες, ορισμένα πράγματα δεν θα είχαν υλοποιηθεί ή θα είχαν υλοποιηθεί με πολύ αργότερο ρυθμό. Αναφέρομαι τώρα στα επιμέρους ε, στοιχεία. Το έγγραφο βέβαια δίνει με λακωνικό τρόπο κάποια παραδείγματα και γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, ζητήσω ε, να δείτε ε, τα πεδία του εγγράφου τα οποία αναφέρουν τα επιτεύγματα, έχουν, μέχρι ποιο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί και τα λοιπά σε αναλυτικό, με αναλυτικό τρόπο. Εδώ θα σας δώσω απλώς κάποια παραδείγματα έτσι ώστε να είναι καλύτερη η απεικόνηση των στοιχείων τα οποία αναφέρονται στο έγγραφο όσον, αφορά ας πούμε το πρώτο, το πρώτο στόχο που είναι η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πούμε ότι εμείς θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε ε, τους ε, οριζόντιους ε, φραγμούς που υπήρχαν μέχρι τώρα, καθώς επίσης και να αντιμετωπίσουμε και να άρωμε και ορισμένους φραγμούς που αφορούν εξειδικευμένα κάποιους τομείς. Στην πρώτη περίπτωση, ας πούμε, μπορεί να είναι οι κρατικές επιδοτήσεις, είναι η αξιολόγηση του περιβάλλοντος επενδύσεων κτλ. Κατά αυτή την έννοια στη Ρουμανία έχουμε ένα ε, επικυρωμένο νομικό πλαίσιο για την πραγματική ε, εφαρμογή του, ε, τον, του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες προμήθειες, καθώς επίσης και μια νέα εθνική υπηρεσία για τις δημόσιες προμήθειες. Έχουν αλλάξει δηλαδή κάποια πράγματα και βλέπουμε ότι και σε άλλες ε, περιπτώσεις ε, και σε άλλες ε, χώρες έχουμε βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων είτε μέσα από την χρήση των αντιστοίχων ταμείων είτε χωρίς. Επίσης, βάση της μελέτης ε, έχει καταδειχθεί ότι οι εκ των προτέρων ε, μπορεί να παίξουν καταλητικό ρόλο ε, σε, στην αλλαγή των, των καταστάσεων, καθώς επίσης μπορεί να παίξουν ρόλο καταλήτη όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στρατηγικής και πολιτικής και να προωθήσουν τις νομοθετικές αλλαγές σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι η υγεία, όπως είναι είναι η εκπαίδευση ε, κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν έχουμε παραδείγματα που βοηθήθηκαν χώρες ε, σε αυτές τις ε, υλοποιήσεις. Το επόμενο στοιχείο ε, είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι έχει υπάρξει επιτάχυνση της, ε, ε, ε, της εφαρμογής και της υλοποίησης του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διευκολύνθηκε από τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων ερεσιμοτήτων τα οποία συνδέονται καθαρά με την υλοποίηση των κανόνων και τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ας πούμε σε περιπτώσεις όπως είναι της Ισπανίας, της Πολωνίας, Πορτογαλίας, ε, έχουμε ε, βοήθεια της και βελτίωση της μεταφοράς των κανόνων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς επίσης και τις οδηγίες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Έχουμε επίσης περιπτώσεις όπως της Κύπρου, της Ισπανίας και της ε, Ιταλίας ε, ε, που αφορούν τον τομέα των αποχετεύσεων καθώς επίσης και την διαχείριση των υδάτων ε, και ε, πρέπει να πω ότι έχουν βοηθηθεί οι χώρες και από εμά και από τις ε, διαχειριστικές αρχές σε πολλούς τομείς έτσι ώστε να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις. Στο σημείο έχουμε το τέταρτο ε, όφελο, το οποίο αφορά την καλύτερη στόχευση της ε, στήριξης ε, από τα ταμεία, αλλά και από άλλες μορφές δημόσιας χρηματοδότησης και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η εφαρμογή των εκτοπροτέρων αριθμοτήτων έχει παίξει υποβοηθητικό ρόλο. Αυτό άλλωστε ε, κατεδείχθηκε στο εργαστήριο ε, που ε, είχατε και εσείς στα τέλη του Νοέμβρη του 2016 ήταν σαφές ότι η παρουσία μιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα πάνω έχει βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο πλαίσιο, να υπάρξουν τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα κριτήρια επιλογής ε, για τα προγράμματα ε, και να οριστούν καλύτερα οι ανάγκες ε, στην κατάρτιση προτεραιοτήτων όσον αφορά τις επενδύσεις. Ε, όσον αφορά το τελευταίο ε, σημείο το οποίο είναι η βελτίωση ε, της διοικητικής ικανότητας και του συντονισμού και εδώ έχουμε πολλές περιπτώσεις των προτέρων ερεσιμότητας που έχουν βοηθήσει στη βελτίωση των θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων των δημοσίων οργάνων και που έχουν βοηθήσει ε, τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην δημόσια διοίκηση ε, και στους εμπλεκόμενους. Έχουμε τέτοια ε, παραδείγματα, σας τα δείχνω στην διαφάνεια, τα οποία ακριβώς απεικονίζουν εν συντομία αυτά τα οποία στο έγγραφο αναφέρονται πολύ καλύτερα. Ας στην Πορτογαλία έχουμε ένα νέο σύστημα μαθητείας και κατάρτισης που αποτελεί τμήμα ενός κυβερνητικού προγράμματος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και αυτό συνδέεται με την εκ των προτέρων με τις και ε, ερεσιμότητες στη Γαλλία, ας πούμε, έχουμε επίσης ε, στα πλαίσια ακριβώς των εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων ε, τοπικούς φορείς που έχουν συμμετάσχει για πρώτη φορά στην προετοιμασία μιας περιφερειακής στρατηγικής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, τώρα ε, βεβαίως υπάρχουν στοιχεία τα οποία περαιτέρω μπορούν να βελτιωθούν. Θα επανέλθω στο επόμενο σκέλος ε, της ε, ε, αναφοράς μου. και σε, στην προκείμενη περίπτωση, ε, όπως και στην προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειξα, ε, το σημαντικό είναι ότι τοπικοί φορείς, ε, περιφερειακοί φορείς έχουν έρθει σε επαφή με την κεντρική κυβέρνηση έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η περιφερειακή συνεργασία. Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο που αφορά τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει, πρέπει να πω ότι εδώ βασιστήκαμε και στην ανάδοση, στο feedback που είχαμε από τους ε, τοπικούς φορείς, από τις ε, ρυθμιστικές ε, και διαχειριστικές αρχές και πρέπει να πω ότι πραγματικά θεωρούμε ότι έχουμε βελτιώσει το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι τοπικοί φορείς και οι επενδύσεις. Όπως όμως υπόθηκε και στο εργαστήριο του Νοεμβρίου, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτό το συγκεκριμένο ε, εργαλείο όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και επομένως ακόμα είμαστε στη διαδικασία ε, της ε, όσον αφορά το ΕΣΥΦ και είναι η πρώτη φορά λοιπόν έλεγα που το χρησιμοποιούμε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, ε, πραγματικά και βάσει των πληροφοριών που έχουμε, έχουμε ε, καλά αποτελέσματα. Επίσης έχουν βελτιωθεί οι συμφωνίες εταιρική συνεργασίας, λαμβάνονται υπόψη νέα κριτήρια. Βεβαίως ευελπιστούμε ότι, ότι θα είχαν ολοκληρωθεί όλα την προηγούμενη χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξέρουμε στο τέλος του καλοκαιριού τι έχει ολοκληρωθεί και τι όχι. Ε, όσον αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής, έχουν ε, ήδη εγκριθεί από τους ε, ε, συνομοθέτες ε, τα βασικά στοιχεία και στην Κομισιόν θεωρούμε, θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Βεβαίως βλέπουμε ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν έχει πάντα εφαρμοστεί σωστά ε, και έχουμε δει ότι ε, επίση ε, και το πεδίο εφαρμογή αλλά και ο αριθμό των εκδομητών ενσωματήτων σε μερικέ περιπτώσει είναι υπερβολικά μεγάλο. Θα πρέπει να το δούμε έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο οι εκδομητών ενσωματήτες μπορούν καλύτερα να προσαρμοστούν στι τοπικέ περιφερειακέ ανάγκε, γιατί αυτή είναι η προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε και βέβαια το ζήτημα είναι κατά πόσον μπορούμε να βελτιώσουμε την καταλληλότητα των προγραμμάτων. Ε, βέβαια, τα... είχαμε και πολύ αξιόλογα σεμινάρια, πολύ παραγωγικά και τα απορίσματά τους ήταν πολύ έγκυρα και πολύ χρήσιμα. Μάλιστα, ένα από τα πράγματα ήταν ότι αυτές οι εκ των προτέρων ε, δεν θα πρέπει να είναι μια, ένα απλό εγχείρημα που ε, κάνουμε τίξ τα κουτάκια. Θα πρέπει να εξακριβώνουμε κατά πόσο έχει επιτευχθεί αυτή η εξάντ, αυτή εκ των προτέρων αιρεσιμότητα και αυτό είναι μια προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τα ωφέλη μια τέτοια συμμόρφωσης ε, τα βιώνουν οι επιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουν οι περιφέρειες, οι εμπλεκόμενες ή τα εμπλεκόμενα κράτη-μέρη την ευθύνη αυτή της προσπάθειας. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει απλώς μια εξακρίβωση και να πούμε ότι okay, ε, πληρείται η αιρεσιμότητα». Μας ενδιαφέρουν τα αυτά ωφέλη που τα νιώθουν τα κράτη και οι περιφέρειες. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουν κτήμα τους αυτή την αιρεσιμότητα. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι η επαρκής διοικητική ικανότητα και συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Είχαμε επαφές με πολλούς ενδιαφερομένους, πολλές με κυβερνητικές οργανώσεις πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες και αυτό είπα και εκείνοι ότι θέλουν μεγαλύτερη συμμετοχή, εμπλοκή και γενικώ είναι ικανοποιημένοι με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα και πιστεύουν ότι απέφερα καρπούς ε, από τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη ανάμειξή του στην όλη διαδικασία. Και το τελικό μας δίδαγμα ήταν η εφαρμογή των προγραμμάτων πριν την υλοποίηση των αρεσιμοτήτων. Ε, κατά κανόνα έχουμε μια τριετή περίοδο χάρη τόσο που γίνονται επενδύσεις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επιδετικά Ταμεία χωρίς ε, πλήρη συνδρομή των ε, ε, προϋποθέσεων με βάση τις αρχές της εκ των προτέρων Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Θα πρέπει να παραμείνει αυτή η τρίτη περίοδο χάριτος. Και τέλος, ε, ένα άλλο θέμα που αναλύθηκε σε αυτό το σεμινάριο ήταν ότι εκπρόσωποι των κρατών μελών είπαν ότι θα πρέπει να ξέρουν εκ των προτέρων εστί τέτοια εκ των προτέρων ερεσιμότητα ώστε να μην επηρεάσει μία σάφιας προς τον ορισμό την ε, επερχόμενη διαδικασία. Ποια είναι τώρα τα επόμενα μας βήματα μετά τη σημερινή συζήτηση και μετά το διαρθρωμένο διάλογο που είχαμε με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις θα κάνουμε την Παρασκευή στο Συμβούλιο μια παρουσίαση του εγγράφου. Και φαντάζομαι θα περιληφθεί και στη συζήτηση του 7ου Φόρουμ για τη Συνοχή τον Ιούνιο, Τέλειο Ιουνίου. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή και τώρα συζήτηση. Υπάρχουν σχόλια, ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε Βανίλη Στερό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στη συζήτηση και μας δίνεται αυτή την ευκαιρία α, ε, μεγαλύτερης ευάθυνσης. Δυστυχώς υπάρχει μια αντίχηση από το μικρόφωνο του ομιλητή. Δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα ακόμη δυστυχώς. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε αυτή την περίοδο για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θέλει να βελτιώσει την νομοθεσία. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές και για τα ΕΣΥΦ, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Παιδωτικά Ταμεία. Και Γι' αυτό και για την καλή εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να ενισχύσουμε την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, που είναι απαραίτητο δομικό υλικό, απαραίτητη προϋπόθεση για, καλύτερη, για καλύτερα αποτελέσματα, για καλύτερες προσεγγίσεις που θα εδράζονται σε αποδείξεις και σε επιδόσεις. Και αυτό είναι το αντικείμενο της παρουσίασης. Πάντως το πλαίσιο προγραμματισμού είναι φταετές και η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων γίνεται στην αρχή με τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, με τα επιχειρησιακά προγράμματα, γίνεται ε, μια εκτίμηση το πόσο αποδοτικά είναι, αλλά τα αποτελέσματα καταμετρούνται πέντε χρόνια μετά, στο τέλος τη περίοδου και έχουμε μάλιστα και ένα παθεματικό, 21 δις, ώστε όσοι έχουν επιδόσεις να λαμβάνουν συμπληρώματα. Και τι γίνεται στο μεταξύ. Έχουμε τρεις εθνικές εκλογές, έχουμε αλλαγές στην πολιτική, στις κυβερνήσεις, στις κυβερνήσεις που έρχονται και παρέρχονται, στη σύνθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ε, μια νεφελώδης κατάσταση λοιπόν. Γι' αυτό και σημαντικό είναι το χρονικό πλαίσιο που εφαρμόζουμε. Γιατί και στις περιφέρειες επειδή θέλουμε επανεκλογή, θέλουμε αυτά αποτελέσματα. Και αν έχουμε τόσο μακροχρόνιες περιόδους ε, ε, εφαρμογής που υπερβαίνουν ε, τον πολιτικό κύκλο και τον εκλογικό, είναι δύσκολο να καταμετρηθούν αυτά τα αποτελέσματα. Πώς λοιπόν αυτό το έργο σας συνδέεται με την προσπάθεια και την πρωτοβουλία του κ. Τίμερμανς για την καλύτερη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είχαμε την έκθεση με βάση το άρθρο 63 και έχουμε τώρα τα βασικά δομικά στοιχεία της περίοδου μετά το 2020 και προετοιμάζουμε και την κοινοβουλευτική αξιολόγηση αυτού του φόρουμ της συνοχής του Ιωνίου και ακριβώς μας προβληματίζουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Συγγνώμη Προϋπολογισμού ζητά περισσότερη, περισσότερο προσανατολισμό και εστίαση στα θέματα ε, αποτελεσμάτων ε, παραγωγής γιατί έχουμε ε, την επίπεδη διακυβέρνηση και έχουμε πολύ αισιόδοξο και πλήρες ε, πλαίσιο και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε καλύτερη νομοθεσία και καλύτερα αποτελέσματα και θέλουμε να πάρουμε καλούς βαθμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα, θα πρέπει να το ξέρουμε θα πρέπει η Επιτροπή Γιούγκερ όταν θα κάνει στο τέλος της τον απολογισμό για το κατά πόσο υλοποίησε την καλύτερη νομοθεσία να είναι σε θέση να εξάγει συμπεράσματα για το αν όντως υπήρξε βελτίωση. Και εμείς ε, οι Ευρωβουλευτές όταν συζητούμε με τους συναδέλφους μας από διάφορες επιτροπές ε, και από εκπροσώπους των νέων εργαλείων του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα πρέπει φυσικά να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια χρονοβόρα διαδικασία όμως που προϋποθέτει πόρους, δυναμικό, που αναμειγνύει και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα από θα ήταν ένα από τα θετικά παραδείγματα του νέου τρόπου και τις νέες μεθοδολογίες εργασίας. Και σε ό,τι αφορά την εκ των προτέρων αρεσιμότητα καταρχήν, μας εξέπληξε που πέρυσι στις συζητήσεις ε, επί τσεχικής προεδρίας ε, στα συμπεράσματα της Πρατισλάβα και της Σλοβακικής προεδρίας μάλλον στα συμπεράσματα της Πρατισλάβα το Συμβούλιο ήταν πολύ θετικό δεν είπαν ότι θα είναι πολύ χρονοβόρα και περιπλοκή διαδικασία, αλλά θέλουν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την πολιτική από κοινού με τους ενδιαφερομένους και να έχουμε κάποιες ενδιάμεσες μεσοπρόθεσμες συμφωνίες για την πολιτική που θα ακολουθήσουν και μετά τα κρατημέλη. Επίσης, πολύ συχνά στην έκθεση μιλάτε για τις ειδικές στάσεις αναχώρα. Αυτό θα είναι σημαντικό μετά το 2020 κατά τη γνώμη μου, ώστε να μπορούν οι χώρες να λαμβάνουν κονδύλια. Και αυτό θα μας ενδιαφέρει και για τη μελλοντική συζήτηση, όχι μόνο για το πώς λειτουργούν τώρα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε στο μέλλον να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και να τις επιταχύνουμε και όλα, να επιταχύνουμε τα αποτελέσματα. Επίσης αναφέρεται τι ε, τις δημόσιες ε, συμβάσεις, κρατικές και άλλα παραδείγματα άλλου τομεί. Υπάρχουν στατιστικά τεκμήρια, όπως αναφέρθηκε στην έκθεση του άρθρου 63, ότι ε, έχουν, αφορούν, 75% όλων των ειδικών συστάσεων ανά και ποιες χώρες ε, απορροφούν κονδύλια και έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γιατί η παρουσίασή σας ε, μου θύμισε μια επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ ε, που παίρνουμε από εδώ και από εκεί διάφορα προϊόντα, τα βάζουμε στο καλάθι μας, στο καρατσάκι μας, αλλά δεν ξέρουμε τελικά τι ψωνίσαμε. Και την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε το πρόγραμμα στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το νέο εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. που ε, προσφέρει επίσης κάποιες δυνατότητε. Ποιες οι διαφορέ όμω μεταξύ αυτού του εργαλείου και των εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων. Είναι σημαντικό ε, με όλα αυτά τα στοιχεία να έχουμε μια πιο περιστατωμένη κρίση κατά το τέλος του περίοδου και να δούμε αν ε, οι εκ των προτέρων αξιολογή, ε, ρεσιμότητες είναι πιο χρήσιμες από το τελευταίο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντως υπάρχει κάποια βελτίωση, αλλά εξακολουθεί να είναι περίπλοκη η κατάσταση για τους ενδιαφερομένους. Και επίσης, ακριβώς επειδή είναι πολύ ευρύς ο χρονικός ορίζοντας ε, και πολύ χρονοβόρο η διαδικασία, δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος τι θα πάει στραβά και τι καλά. Ευχαριστώ κύριε Βαμίλτον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκράντ για την πολύ καλή παρουσίαση. Ούτε καν το πίστευα διαβάζοντα για την προσθέμενη αξία των εκ προτέρων αιρεσιμοτήτων. Ακριβώ για αυτά που είπε και ο συνάδελφο ε, ε, ο Λάμπερτ. Στη ε, σελίδα 18 λέτε ότι χρήσιμο θα ήταν να δούμε το δεχόμενο θετικών κινήτρων πέραν της αναστολής πληρωμών αν χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Το είπε και ο Λάμπερτ. Υπάρχει πρόβλημα με τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα κίνητρο ή έχετε άλλες ιδέες που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ήδη από τώρα. Θα ήταν κάτι πιο θετικό από την αναστολή πληρωμών απλά. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι ορισμένες από τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, άρα το να απειλείται με αναστολή πληρωμού δεν είναι η μόνη απάντηση. Το ερώτημά μου δηλαδή είναι ποιες είναι οι άλλες επιλογές σας, ιδίως ε, σε σχέση και με τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα που θα συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ η κυρία έτσι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για εκ των προτέρων αρισιμότητες, Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε τι θέλουμε να πετύχουμε σε επίπεδο κρατών μελών με αυτές τις αρεσιμότητες. Αυτό το ε, συντελεστή έκπληξη θα πρέπει να τον περιορίσουμε όταν μιλάμε ε, για τις εκ των προτέρων αρεσιμότητες που από τα κράτη-μέλη, διότι αυτό βασικά πρέπει να λέγεται στην αρχή, να το περιλαμβάνει ο κανονισμός και να είναι ξεκάθαρο για τα κράτη-μέλη τα θέλουν να επενδύσουν στην ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην υγεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στις μεταφορές, σε οποιοδήποτε κλάδο, ότι θα πρέπει να έχουν στρατηγικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρουν ε, το που βρίσκονται, το ότι θέλουν να πετύχουν και πώς συνεισφέρουν τα κονδύλια την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτεύξη των στόχων αυτών. Δεν πρέπει ουσιαστικά να είναι και κάτι πιο τόσο πολύπλοκο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την περίοδο, 2014-2020, είναι πολύπλοκα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν κρεμεί ε, των προτέρων ερεσιμότητες ε, και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα και συμφωνώ με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή καταρχάς τι θα κάνουμε με τις των προτέρων αρισιμότητες που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, εκπληρωθεί και δεν ξέρω αν θα ήταν δυνατόν οι χώρες να έχουν με κάποιο διαφορετικό τρόπο να δείξουν τι θα πετύχουν, δηλαδή και χωρίς τα έγγραφα αυτά, τα οποία χρειάζονται βεβαίως ε, εκ προτέρων, έγγραφα εκ των προτέρων αρισιμότητας, αλλά μήπως έχουν κάποιον άλλο τρόπο να δείξουν τι θα κάνουν, να γίνει μια εντελεχής ανάλυση και έπειτα να αντιληφθούν διδάγματα για το μέλλον. Άρα θα θέλαμε οι εκ των προτέρων αρισιμότητες να περιγράφονται πιο γενικά, ώστε να ξέρουν από τον προτέρων οι χώρες τι πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να δαπανίσουν πόρους για τους συγκεκριμένους τομείς και να χρησιμοποιήσουν για αυτούς τους στόχους, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος, δεν βλέπω να θέλει κάποιος. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα και νταμάτο έχει το λόγο. No problem. Um, solo una, una Μια ερώτηση στην Κομισιόν μόνο. Θα ήθελα να μας πει δύο λόγια παραπάνω σχετικά με ενδεχόμενες προόδους όσον αφορά τις ε, κρατικές επιδοτήσεις ε, και όσον αφορά και τα δημόσια, τις δημόσιες προμήθειες ε, για όλες τις χώρες αλλά ιδιαίτερα για την Ιταλία αν είναι δυνατόν. Ε, και επίσης ε, θα ήθελα να μας πει δύο λόγια σχετικά ε, με τα ειδικά, τα ειδικά σχόλια για το 2014 όσον αφορά ακριβώς τις δημόσιες προμήθειες και τις διαδικασίες αυτές στα πλαίσια των δικών ταμείων. Ευχαριστώ. Αν μπορείτε να απαντήσετε, λέει πρόεδρος, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Βανίστελ Ρόι Νομίζω ότι μιλήσατε πολύ για το timing, για την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής. Και νομίζω ότι ένας από τους βασικούς στόχους ε, των ταμείων ΕΣΥΦ ε, είναι να βρουν κονδύλια για, μικρο, για δομικές και μακρο, μάλλον βράχοι μεσοπρόθεσμες επενδύσεις. Έχουμε τους ετήσιους προπολογισμούς ε, που παρέχουν σταθερότητα στους καιρούς αυτούς για επενδύσεις στα κράτη-μέλη. σε ό,τι την καλύτερη νομοθεσία. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον κύριο Τίμερμανς δηλαδή, γενικά για την καλύτερη νομοθεσία. Και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα REFIT και στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση των ε, συνθηκών για τους δικαιούχους. πάντα σε σχέση με την καλύτερη νομοθεσία. Νομίζουμε ότι κάνουμε κάποια πράγματα και ήδη υπάρχουν και σχετικέ προτάσεις στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus. Πολλά δε προέρχονται από την απλούστευση των κανόνων. Μετά από τα συμπεράσματα τη ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλούστευση. Και το έργο αυτής της ομάδας συνεχίζεται και φέτος εξετάζουν τη βελτίωση της νομοθεσίας για τη νέα περίοδο. Αυτή είναι η εντολή τους. Διακόπτει ο κ. Βανίστελ Ρόι. Εσείς δουλεύετε με όλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάξει. Όμως το δικό μου ερώτημα είναι, τη μέθοδο εργασίας μας ε, την εκτιμούν δεν υπάρχει άλλος τομέα πολιτική που να μελετά τόσο εντελεχώ όλα τα σημεία. Θέλετε να έχετε μαθηματικούς τύπους και τα λοιπά για όλα. Είναι πολύπλοκο. Τι λένε, ναι, είναι ένα σύστημα ή λένε όχι, είναι πολύ δυσκίνητο, δυσανάλογο, πολύπλοκο κτλ. Μπορείτε να μας δώσετε το μέσα στην απάντησή σας για την ουσία του ζητήματος, για το ψητό. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, γενικά ε, ασχολείται με έναν περιπολισμό προσανατολισμένο πιο πολύ στα αποτελέσματα, άρα βλέπω μια πραγματική μετατόπιση. Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε, αλλά... Δεν μπορώ να κρίνω ε, και ελπίζω να είναι θετικό ο τρόπος που βλέπουν το έργο σας πάνω στον κανονισμό ΕΣΥ. Και θα δούμε τι θα γίνει για, τον επόμενο, ε, για την επόμενη περίοδο που θέλουμε να έχουμε ένα πολύ πιο εύρωστο, ε, μάλλον ε, στέρεο σύστημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση της Κομισιόν. Δεν μπορώ να μιλήσω όμως εγώ σαν των κεντρικών υπηρεσιών. ελπίζω να είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά δεν μπορώ να σας πω. Αλλά νομίζω ότι και η δική μου γαμαδέλτα θεωρεί Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, αλλά είναι ένα στέρεο ε, σύστημα προσαρτησμένο στα αποτελέσματα και αν το βάλουμε μαζί και με τι ε, ρεσιμότητε, πραγματικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, σοβαρέ επενδύσει ε, και αποτελέσματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προπολογισμού και ιδίω στο πολιτικό πλαίσιο που έχουμε σήμερα με όλε αυτέ τι αμφισβητήσει. Δεν μπορώ από πέραν τούτου κάτι ακόμη όμω. Ευχαριστώ. Επόμενο δεύτερο σημείο για την Τσεχική Προεδρία. Ήταν θετική. Δεν ξέρω αν κάνετε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό. Οι περισσότερε συνεισφορέ που πήραμε ω feedback είναι ότι το προτέρων οι απέδωσαν. Και στο διαφανή διάλογο με του εμπλεκόμενου φορεί ε, ακούμε πολύ θετικά σχόλια σε σχέση με τι αιρεσιμότητε αυτές. υπήρξαν ε, προβλήματα κατά το παρελθόν, δεν μετακινήθηκαν, ε, δεν άλλαξαν κάποια πράγματα που όμως τώρα μπορούσαν να αλλάξουν χάρη σε αυτές τις εκ των προτέρων ρεσιμότητες. Άρα είναι θετικό ε, το feedback που έχουμε από τις αρχές και σε ό,τι αφορά το workshop που αναφέρατε. Μπορεί να μην είναι 100% όλες τις περιφέρειες και όλα τα κρατημέλη υπέρ, η μεγάλη πλειοψηφία όμως είναι. Το τρίτο ε, στοιχείο, το οποίο αφορά τις συστάσεις αναχώρα, ειδικέ τάσει αναχώρα, ε, αναφέρεται σε μία μελέτη, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι μία μελέτη η οποία ακριβώς αφορά τον, τον αντίκτυπο που έχουν ε, τα ταμεία, το Ταμείο Επενδύσεων και διαφορετικά επενδυτικά ταμεία σε σχέση και με τις ε, συστάσεις ε, αναχώρα. Ε, ε, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει προχωρήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως δεν μπορώ να σας δώσω ε, στοιχεία συγκεκριμένα. Τώρα, όσον αφορά το... Η SRSS και το τι μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, ε, εμείς ε, συζητούμε στο έγγραφο τα διδάγματα του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία στρέφεται περισσότερο ε, προς το μέλλον όσον αφορά δηλαδή, την υπηρεσία στήριξη διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Και όσον αφορά τα στρατηγικά έγγραφα, να σας πω ότι όντως αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της μελέτης. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί. Γνωρίζουμε ότι 86% έχουν καλυφθεί ε, και έχουν αλληλεθεί από την Κομισιόν, αλλά παραμένουν ε, ε, ε, επίσης ε, και 40% που δεν έχουν ακόμα κατατεθεί. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν εάν έχουν καλυφθεί οι προϋποθέσεις ή όχι. Η Κομισιόν το 12 ήδη είχε κάνει ένα προσχέδιο. Από την πλευρά της Κομισιόν λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν όλο τον απαραίτητο χρόνο έτσι ώστε να ε, ολοκληρώσουν τις ε, ε, προϋποθέσεις. Ξέρουμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα σε ορισμένες χώρες, άλλες τα κατάφεραν, άλλες όχι, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό το Staff Working Document θέλει να δείξει ποια είναι η θέση της Κομισιόν, ποια είναι η γενική κατάσταση, αλλά βεβαίως δεν αποτελεί τελική ανάλυση. Επίσης, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα ε, πολύ καλά αυτό που με ρωτήσατε όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Ρωτώ ε, λοιπόν και σας ξαναρωτώ εάν η Κομισιόν έχει ήδη αποτελέσματα όσον ε, αφορά ε, τις εκτοπροτέρων ερεσιμότητες, όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, public procurements, για όλες τις χώρες και ιδιαίτερα για την Ιταλία. to Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Εάν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, ε, ε, πρέπει να σας πω ότι ε, έχουν αναλυφθεί δράσεις σε ορισμένες χώρες, σε πολλές χώρες όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και τις εκ των προτέρων Μάλιστα αναφέραμε και μερικά από τα επιτεύγματα στις διαφάνειες στην εργασία. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείται αποτελέσματα Όταν ένα κράτο μέλος αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί μια εκ των προτέρων ερεσιμότητα, εμείς ελέγχουμε με τις αρμόδιες αρχές της ε, Κομισιόν ε, εάν πραγματικά έχει ολοκληρωθεί ε, η εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Τέσσερις χώρες ε, δεν έχουν ακόμα ε, δώσει ε, τα τελικά στοιχεία όσον αφορά τις εκ των προτέρων ερασιμότητες για τις δημόσιες προμήθειες. Δεν ξέρω να απαντώ στην ερώτησή σας. Okay. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Επομένως, ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, παρουσίαση του εγγράφου και σας ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα του τέταρτου φόρουμ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το τέταρτο φόρουμ για τις εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές και την προσπάθεια για μια ανανεωμένη στρατηγική έλαβε χώρα υπό την αιγύδα της Κομισιόν στις 30 και 31 Μαρτίου του 2017 το πρόγραμμα ε, το έχετε σε ηλεκτρονική ε, μορφή και επίσης ε, έχετε και όλα τα έγγραφα και τις παρουσιάσεις ε, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Αποτέλεσε μια καλή πλατφόρμα ε, συζήτησης και επαφής μεταξύ των απόκεντρων περιοχών από τη μία πλευρά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ε, ευρωπαϊκά όργανα και ε, ε, υπηρεσίες από την άλλη πλευρά. Έγινε αναφορά στην νέα στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κυρίως όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, ε, στα πλαίσια της αναθεώρησης στρατηγικής της ε, Επιτροπής, ε, η Κομισιό μας αποφάσισε να συγγράψει έκθεση, βάσει του άρθρου 349 ακριβώς με θέμα τη στρατηγική της απόκεντρες περιοχές. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση στην συνεδρίασή μας του μηνός Μαΐου. Η έκθεση αυτή ε, θα καταγράφει την θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση. Επομένως είναι ιδιαίτερος επίκαιρη η συζήτηση η σημερινή, λαμβάνοντα υπόψη ότι θα πρέπει να συζητηθεί και η έκθεση. Ε, καλούμε τους εκπροσώπους λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους έχουμε εδώ, ναι, να πάρουν το λόγο. Και θα σας δώσω το λόγο λοιπόν αγαπητή κυρία. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Αυτή η τέταρτη ε, ε, διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουμ ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και αντανακλά την πολύ αγαστή εταιρική σχέση που έχουμε με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, τις περιφέρειες, τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από πολλούς ευρωβουλευτές. Ήταν και ο κύριος Ομαρτζή, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές. Γενικώ είχαμε 658 συμμετέχοντες σε αυτή την ε, διοργάνωση, 700 ε, το παρακολούθησαν μέσω του του διαδικτύου, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον αυτή, για αυτή την εκδήλωση. Επίσης είχαμε 232 προσώπους από περιοχές, ε, τόσο από εθνικούς ε, ε, φορείς, 150 από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και 50 δημοσιογράφους που κάλυψαν αυτό, αυτή την εκδήλωση ήταν εκτενής ε, και πολύ αξιόλογη η κάλυψη, κάτι που αντικατοπτρίζει, επαναλαμβάνω, την πολύ εργαστή συνεργασία που έχουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. που έλαβε μέρος, όπως σας είπα, σε πολλά μέρη του προγράμματος, στην εισαγωγή, ε, που ένα μήνυμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μέσω βίντεο και είχαμε και πρωινές και απογευματινές συνεδριάσεις και επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές και τους βοηθούς και συνεργάτες τους που μας βοήθησαν στην προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης. Βρισκόμαστε στην απαρχή βέβαια της διαδικασίας και θα είναι χρήσιμη συζήτηση για να τροφοδοτήσει την ανακοίνωση που θα υποβάλουμε στα τέλη του έτους και που θα ανανεώσει την στρατηγική μας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ε, ήταν παρόν στην εκδήλωση και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπενθύμησε ότι σε ό,τι αφορά αυτή την ε, ανανέωση της στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, ε, θα ήθελε η νέα ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι καινοτόμα, φιλόδοξη. Ανέφερε τα μέχρι, τις μέχρι τώρα προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικώς σε από απόκεντρες περιοχές και τα αποτελέσματα που απέφεραν. Ε, και ανέφερε τα ενδιαφέροντα ζητήματα και μάλιστα εν και της κρίσης που είχαμε στη Γουιάννα αναφέρθηκε αυτό στη διάρκεια της εκδήλωσης, που ευτυχώς τελικά είχε αίσια έκβαση, παρά τις αναταραχές. Σίγουρα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση που μας στείλετε από την Επιτροπή σας για την εφαρμογή του άρθρου 349 και προσβλέπουμε σε πολύ στενή συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί και η έκθεσή σας, επαναλαμβάνω, θα επηρεάσει ε, το περιεχόμενο της ανανεωμένης μας στρατηγικής για τις εξόχως απόλυτες περιοχές. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, μήπως. Ο κύριος ε, Μέντσεμπορκ. Μια γενική ερώτηση. Ε, ε, ζητήσαμε πιο ε, έντονη εφαρμογή του άρθρου 349, όπως επισήμανε και ο κ. Σομαρτζέ στην εκδήλωση. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ζήτησαν κάτι τέτοιο στην, στο φόρουμ αυτό. Και εσείς τι γνώμη έχετε, γιατί θεωρώ ότι για την έκθεση ο Μαρτζή και τη σχετική έκκληση που απευθύνουμε εκεί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Υπήρχε αντίστοιχο αίτημα των και απόκεντρων περιοχών για πιο εντατική εφαρμογή του άρθρου 349. Ο κύριος ε, Μάνσκου. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διοργάνωση αυτού του τέταρτου φόρουμ που έλαβε χώρα πριν από λίγες εβδομάδες, σχετικά πρόσφατα. Και μάλιστα χαιρετίζω την ε, εκπροσώπηση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, γιατί ήταν παρούσα και η Επίτροπο Κρέτσου, η αρμόδια Επίτροπο, αλλά και ο ίδιο ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Γιούνκερ. Κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και την ευαισθησία τη ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Οι ιδιαιτερότητε αυτών των εξόχων απόκεντρων περιοχών και των ε, υπερπόντιδων διαμερισμάτων και τα προβλήματά του είναι γνωστά. Και μάλιστα η κατάσταση στη Γουιάννα ακριβώ που μα ε, δείχνει τα δεινά και τα χάντικα, τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ε, προβλήματα που αφορούν την υποδομή, την υγεία, την παιδεία ε, ή την έλλειψη οικονομικών προοπτικών, μεταξύ άλλων. Και εδώ και χρόνια βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας συμπαρίσταται, αλλά Λυπάμαι που στο φόρουμ αυτό, σε αυτό το τέταρτο φόρουμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσε την ε, αίσθηση ότι θέλει να εφαρμόσει πλήρως το άρθρο 349 και κυρίως ε, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή του άρθρου 349 και που ε, δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, να λάβουν ε, εξαιρέσεις. Και μάλιστα χάρη σε αυτή την ομολογία δίνεται λύση σε μία, μία, μία φιλονική που υπήρξε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερμηνεία του άρθρου 349. Δεν θα μπορούσε λοιπόν με βάση την τελευταία νομο, νομολογία του ΔΕΚ να υποβάλει προτάσεις για εξαιρέσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών από, το, από κάποια διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και των συνθηκών. Και οι ερετοί εκπρόσωποι των εξόχων απόκεντρων περιοχών αλλά και εκπρόσωποι φορέων από τις περιοχές αυτές είχαν συγκεκριμένα αιτήματα και είχαν την αίσθηση μερικές φορές ότι ήταν χαμένη η ευκαιρία αυτό το φόρουμ γιατί δεν ένιωσαν μεγάλη ανταπόκριση ως προς τα αιτήματά τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θεώρησαν ότι αφογκράστηκε ε, τα αιτήματά τους. Ε, βέβαια, απουσιάζει ο εισηγητή τη έκθεση, ο κύριο Μαρτζή, αλλά θα ήθελα να την υπόψη την έκθεσή του για την καλύτερη εφαρμογή και την πιο έντονη εφαρμογή του άρθρου 349 τη συνθήκη, ώστε να μπορέσουμε και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεταφέρουμε ε, και να γίνουν ακουστές οι πολυάριθμες ε, ε, τα πολυάριθμα αιτήματα των εξόχων απόκεντρων περιοχών. Και επαναλαμβάνω, λάβετε υπόψη την τελευταία απόφαση του 10 για τα δικαιώματα αυτών των εξόχων απόκεντρων περιοχών, προκειμένου να εφαρμόσετε αντίστοιχα το άρθρο 349 και να επιτρέψετε χάρη σε εξαιρέσει στι ε, περιοχές αυτές ε, να απολαύσουν και αυτέ μια αρμονική ανάπτυξη δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ήταν πολύ σκληρές αυτές οι διαταραχές ε, στην Γουιάννα που κράτησαν ένα μήνα ολόκληρο και μάλιστα έμεινε όμοιρη αυτή η περιοχή για ένα μήνα και επλήγει ιδιαίτερος από τα φοβερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως ε, τέτοιες απόκεντρες περιοχές. Κύριε Τσέλερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όποιοι με γνωρίζουν θα ξέρουν ότι φυσικά και σε ό,τι αφορά ιδίω ε, τι άκρω ε, απόκεντρε περιφέρειε. Ε, είμαι υπέρ τη ανάληψη δράση και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να την χείρα βοηθεία σε αυτές τις περιφέρειες, να σταθεί στο πλευρό τους. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τις απόψεις που ακούσαμε πρόσφατα από τους εκπροσώπους των ε, από απότερων περιφερειών, πρέπει να πω ότι όλες αυτές ανήκουν σε ένα κράτος μέλος και άρα αυτό το κράτος μέλος έχει τις περισσότερες ευθύνες, τις ευθύνες μάλλον εξ ολοκλήρου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μειώσει τις ανισότητες ε, και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, τα δέοντα ώστε τα μειονεκτήματα και οι ανισότητες να περιοριστούν, να παράσχει δηλαδή ενίσχυση ως προς αυτό. Και ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν ε, περιφέρειες εκτός ε, της ε, υπηρετικής Ευρώπης και που ανήκουν σε άλλες υπήρους, αυτό πρέπει να θεωρηθεί πλεονέκτημα και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες από αυτές τις υπήρους που θέλουμε να ενισχύσουμε σε σχέση με ό,τι είχαμε κάνει στο παρελθόν. και επειδή υπάρχουν κάποιοι γεωγραφικοί περιορισμοί, ε, δεν υπάρχουν ε, ανοιχτά ε, σύνορα, ιδίως ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες αυτών των εξόχως από και των Πρέπει λοιπόν να απλωστεύσουμε τα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα και αυτό είναι μια απέτηση την οποία πρέπει να φέρει σε πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος υπάρχουν Άλλοι συνάδελφοι θα ήθελαν το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπουρντή θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να σας επενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο φόρουμ ήταν μια δημόσια συζήτηση. Είναι δηλαδή για την Κομισιόν ώρα να ακούσει ε, και με βάση τις προτάσεις θα καταθέσει εν συνεχεία τις ε, δικές της προτάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ε, στρατηγικής, ανανεωμένης στρατηγικής που θα συζητηθεί. Αυτό το φόρουμ που διοργανώθηκε είχε ως στόχο όμως όπως πάνω να ακούσουμε, να γίνει μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια εμείς να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τα στήματα που ετέθησαν. Ε, για να επαναλάβω κάτι που ανέφερε ο κύριος Μανσκούρ ε, για την, μια εκδήλωση πολύ ψηλού επίπεδου που είπε ότι ήταν αυτό το φόρουμ πράγματι εκπροσωπήθηκε σε ύψη του Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι υπενθύμησαν αυτή την ομολογία, αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Ε, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε μάλιστα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ. Άρα στο ανώτατο επίπεδο της Κομισιόν είναι γνωστό το θέμα και το προσέχουμε ιδιαίτερος. Επίσης σημαντικό είναι, ε, στην έκθεση του κ. Μαρζή που δεν έχει εγκριθεί ακόμη βέβαια, να διατυπωθούν προτάσεις ε, για τη μελλοντική αυτή ανακοίνωση. Σε ό,τι είπε ο κύριος ε, Τσέλερ, δεν νομίζω ότι πρέπει να τα περιμένουμε όλα από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές πολιτικές και στο περιθώριο του φόρουμ είχαμε ομάδες υπερογνωμόνων που συζήτησαν σημαντικά ζητήματα για τις εξόδους από κεντρές περιφέρειες, πράσινη και κυκλική οικονομία για παράδειγμα, η ψηφιακή πρόσβαση, οι μεταφορές. Όταν λοιπόν με τους εμπειρογνώμονες από αυτές τις περιφέρειες ε, εξετάζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι αυτή που πάντα ε, δημιουργεί εμπόδια, αλλά και τα εθνικά κράτη. Οι εθνικέ νομοθεσίε δεν επέτρεψαν ενδεχομένω κατά ανάγκη την απαιτούμενη ευελιξία στι εξόδου από κεντρέ περιφέρειε για να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματά του. Ε, και πραγματικά ε, θα πρέπει να ε, μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και τόσο πλούσια εταιρική σχέση με αυτές τις περιφέρειες, ε, γιατί κάθε χώρα έχει ε, τα δικά της πλονεκτήματα, είναι, έχει το δικό της πλούτο. Όλες οι προτάσεις ε, που διατυπώθηκαν μέσω του μνημονίου της 31ης διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο Γιούγκερ. Ένα πολύ σημαντικό έγγραφο είναι αυτό, που έρχεται να συμπληρώσει την έκθεση του Κοινοβουλίου το αναλύουμε και αυτό το έγγραφο ε, εντελεχέστατα με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Και όλες οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί και στο πλαίσιο τη συζήτηση μεταξύ πολιτών αναλύονται από τι υπηρεσίε Κομισιόν για να δούμε πώ μπορούμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Η ανακοίνωση θα εγκριθεί πριν τη συζήτηση για τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικές Φυσικά και δεν θέλουμε να προεξοφλήσουμε τι συζητήσει για τι νέε δημοσιονομικέ προπτικέ στην ανακοίνωση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά καινοφανή στοιχεία και νέοι ελπιδοφόροι ε, τομεί και θα πρέπει εκεί να δώσουμε την ε, έμφαση. Και όπω είπε και ο ίδιο ο πρόεδρο Γιούνκερ, αληθεύει, το υπενθύμησαν άλλωστε στην προηγούμενη συζήτηση στην Επιτροπή Ρέγγι η συναδελφοί σα και κύριο Σομαρζή ότι υπάρχουν πολιτικέ που έχουμε λίγα ειδικά μέτρα μέχρι στιγμή. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, και αυτό κάνουν με τι ε, αρμόδιε υπηρεσίε, θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα στι από κέντρε περιφέρειε. Να μην τι ξεχάσουμε. Να μην τι αφήσουμε κατά μέρο. Και αυτό στο δυνατόν νωρίτερα, ανάντι. Όχι δηλαδή να θεραπεύσουμε, καλό το προλαμβάνει του θεραπεύν λέμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Και όχι εκ των υστέρων να ερχόμαστε να διορθώνουμε τα πράγματα και αυτό να είναι και πιο προβληματικό ενίοτε. Τέλος, θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το είπατε κιόλας, υπήρξε το θέμα τη απλούστευσης. Ήταν πολύ σημαντικό ζήτημα. Μιλάμε για την πραγματική απλούστευση που μπορούμε να έχουμε για τα προγράμματα μετά το 2020. Γιατί για αυτές τι περιφέρειες η συσσόρευση διαδικασιών δημιουργεί μεγάλο άχθος ε, πολλές φορές και δυσκολεύει τους δικαιούχους. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ολοκληρώνουμε το συζήτηση. τη συζήτηση για το σημείο αυτό. Πάμε με ηλικιώδη ταχύτητα σήμερα το απόγευμα. Και έτσι ολοκληρώνουμε και το, τη δημόσια μας συνεδρίαση. Και ρωτώ τους συντονιστές αν είναι έτοιμοι να συνεχίσουμε αμέσως μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Να μην ε, περιμένουμε. Πολύ ωραία. Οπότε ολοκληρώνεται το δημόσιο τμήμα της συνεδρίας και παρακαλώ όσοι δεν είναι συντονιστές να εγκαταλείψουν την αίθουσα.